Κυρίες, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας καλωσορίζω, αυτούς που είναι εδώ τουλάχιστον. σε πιο γρήγορα αρχίσουμε, τόσο λίγο θα τελειώσουμε. Θα ήθελα να εγκρίνετε την μισή διάταξη, δηλαδή να αλλάξουμε τη σειρά του 3 και του 4. Δεν ξέρω γιατί, για κάποιους λόγους, τέλος πάντων. Και στις ψηφοφορίες, η ψηφοφορία 9 θα γίνει πρώτη Και στο σημείο 11 η Υπουργό ε, Κριστίνα Καρμέλια θα αντικαταστεί από τον, Υφυπουργό, από τον Υφυπουργό. Αυτό δεν είναι κάτι που θα αποφασίσουμε, έτσι κάνουν αυτή τι να κάνουμε. Λοιπόν, αν συμφωνείτε, εγκρίνουμε την μεσαία διάταξη με τεράστιε αυτέ τι αλλαγέ που σα προανήγγειλα και θα αναπαράσουμε στο σημείο 3 τη μεσαία διάταξη αυτό που ήταν παλιά δηλαδή. Ενδυνάμωση χημικό, βιολογικό, ρεδιολογικό και πυρηνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόγραμμα CBRN, εκεί γνωμοδοτούν και ο συνάδελφος Φράνκο είναι αρμόδιος. Και ήθελα να δώσω το λόγο λοιπόν, να διαφωνείτε. Παρακαλώ. Je Σας υπενθυμίζω ότι οι διατάξει για θέματα εσωτερική ε, ασφάλεια και φυσική προστασία είναι θέμα των αρμοδιότητων κρατών μελών. Αλλά μια συνεργασία και εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται ότι είναι από την άλλη μεριά ουσιαστική. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράση στον τομέα τη χημική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική ασφάλεια που είναι γνωστό CBRN είναι κύρια πρόοδος ε, μετά από την τρομοκρατική δράση της 11 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος στόχος της δέσμης μέτρων που αποτελούν το πρόγραμμα δράσης CBRN μια εκατοντάδα περίπου μέτρα, είναι να υποστηριχτούν οι προσπάσεις που καταβάλλονται σε όλα τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό της ασφάλειας και να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων. Το παλάκι είναι ήδη στο γήπεδο των κρατών μελών και εμείς ως ευρωβουλευτές θα πρέπει να τους ε, κινητοποιήσουμε να εφαρμόσουν γλίγορα και αποτελεσματικά αυτό το σχέδιο. Ένας χρόνος πέρασε από την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 24 Ιουνίου 2009 και είναι πολύ ένα χρόνο. χωρίς ισχυρό πολιτικό μήνυμα από σκοπιά μα. Η δυνατότητα σήμερα τα όπλα μαζικής καταστροφής να πέσουν σε χέρια των δημοκρατών είναι η μεγαλύτερη απειλή της ασφάλειας που έζησε ποτέ η Ευρώπη. Παρόλο που δεν έτυχε ποτέ θύμα επιθέσεων CBRN η Ευρώπη σε μεγάλη κλίμακα, παρόλα αυτά πρέπει να περιμένουμε το χειρότερο. Η κατασκευή μιας βόμβας ε, αυτού του τύπου θα μπορούσε να πλήξει τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Θυμάστε τις επιθέσεις με άντραξ ή τις επιθέσεις ε, με το αέριο Σαρίν στο μετρό του Τόκιο. Θα πρέπει λοιπόν να δειχθούμε υπεύθυνοι συνετή, αποτελεσματική. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης προτείνει μία ε, σφαιρική προσέγγιση βασιζόμενη σε τρία τμήματα της ίδιας αλυσίδας. Πρόληψη, ανείχνευση και αντίδραση. Αυτοί οι τρεις άξονες της ε, εργασίας θα πρέπει να μας ε, κινήσουν. Δηλαδή πολιτική βούληση, εφαρμογή μέτρων και έρευνα. Εγώ θα ήθελα καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τις προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση προτύπων κατά της διάδοσης για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη διεύρυνση των ε, πυρηνικών και ραδιολογικών όπλων και να προστατευτούμε επίσης από βιολογικά και χημικά όπλα. στη γνωμοδότησή μου καλό για μια ευφυή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ορισμένε χώρε είναι πιο προχωρημένε από τι άλλε στον τομέα τη ασφάλεια CBRN. Καλύτερα λοιπόν, αντί να επικαλύψουμε τις προσπάθειε να δράσουμε σκόρπια, ας ανοίξουμε τα εργαστήριά μας, ας ενώσουμε τις προσπάθειες και τις ικανότητές μας. Είναι πια καιρός να υπάρχει μια πραγματική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική στον τομέα της αστικής ασφάλειας με μια διαδικασία ε, έγκρισης των διαδικασιών και των εξοπλισμών. Πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στην ΣΥΠΑ στην Κίνα γιατί αυτές οι χώρες έχουν πολύ αυστηρά κριτήρια που οι επιχειρήσεις μας δεν μπορούν να σου. Ας κάνουμε το ίδιο κι εμείς. Να μην χάνει τη βιομηχανία μας σε αντιπαραγωγικές ε, διατάξεις. Επίσης, προτού ξεκινήσουμε νέα προγράμματα ακριβά έρευνας, ας εξετάσουμε την απόδοση της ισχύουσας ε, τεχνολογίας και ας αξιολογήσουμε καλύτερα τα ε, προγράμματα επίδειξης και τη διάθεση των σχεδίων αυτών στην αγορά. Τέλος, λέω, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη στρατηγική συνεργασία και μεταξύ μας και με εταίρους σε διεθνές επίπεδο. Αγαπητοί συναδελφοί, περιμένω με υποσημισία να ακούσω τις απόψεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Äh, Σα ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Ένσου, ο σκιός ηγητής, ε, έχει το λόγο από τους, Σοσιαλιστέ. Ε, σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω είπατε, είμαι σκιώδη ηγητής για την έκθεση αυτή από του Σοσιαλιστέ και δημοκράτε. και είχα την ιδιαίτερη χαρά να συνεργαστώ με τον συνάδελφο Γκάστον Φράγκο που είναι ο βασικός εισηγητής, αλλά είχα συνομιλήσει και με τους υπόλοιπους συναδέλφους που ενδιαφέρθηκαν για το θέμα αυτό. Υπήρξαν δύο στάδια στη διαδικασία ρύθμισης και συντονισμού των δραστηριοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί το CBRN. Ε, πάει ένας χρόνος που μας υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανακοίνωσή της και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχουν λάβει ε, τα απαραίτητα μέτρα, αλλά βρισκόμαστε σε πρωταρχικό στάδιο της εφαρμογής. Περιμένουμε μια έκθεση της διαδικασίας εφαρμογής που θα υποβάλει το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, ε, η κατάσταση μας έδειξε ότι υπάρχουν και μερικοί κάποιες ε, απρόσμενες, απροσδόκητες καταστάσεις. Είχαμε την πετρελοκυλίδα στο Μεξικό, είχαμε τη γρήπη H1N1, είχαμε το σεισμό στην Αϊτή, αστάθμητοι παράγοντες και ανωτέρα βία. Γι' αυτό, επειδή υπάρχουν τις κατεπίγουσες ε, περιστάσεις, θα πρέπει να έχουμε προβλέψει ένα μηχανισμό άμεσης αντίδρασης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα και να περιορίσουμε τις αρνητικές τους συνέπειες. Όπως είπε και ο συνάδελφος ε, Φράνκο Γκαστόν, έχουμε πολλά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τα προϊόντα χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας. Θα πρέπει με ευφύ τρόπο να αποτρέψουμε για να αντιμετωπίσουμε απειλές από τρομοκρατικές ομάδες. Η χρηματοδότηση της έρευνας αυτής μπορεί να γίνει μέσα στα πλαίσια του 7ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου, όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Ταυτόχρονα θεωρώ πολύ σημαντικό για να προλάβουμε τρομοκρατικές ενέργειες ε, με τη χρήση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών όπλων, να διαμορφώσουμε μια βάση δεδομένων όλες τις ουσίες που εμπίπτουν ε, ε, σε αυτή την κατηγορία χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών ουσιών και να αποφύγουμε το λαθρεμπόριο τέτοιων ε, επικίνδυνων ουσιών. Επίσης, ε, πρέπει να δούμε ποιες τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποιούν τέτοια όπλα, χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά ή πυρηνικά. Και νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δυνατότητες του διαδικτύου προκειμένου να διαδώσουμε στους πολίτες κάποιες βέλτιστες πρακτικές για μέτρα ασφάλειας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Θα πρέπει να αποφύγουμε παράνομη διακίνηση πληροφοριών για ουσίες χημικές, ραδιολογικές, βιολογικές και πυρηνικές. Θα πρέπει επίσης να ενημερωνόμαστε για όλες τις φάσεις της έρευνας ε, για τέτοια ζητήματα και να ενημερωνόμαστε με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνα. Η χρήση προϊόντων CBRN είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση, να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και με υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση σε στενή φυσικά συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Πολ Ρούμπιχ. Σας ευχαριστώ. Hm, äh, äh, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή γιατί πραγματικά η ασφάλεια για μας είναι πολύ σημαντική και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιλέξει το σωστό τρόπο και τη σωστή διαδικασία για να βελτιώσει την κατάσταση διαδίδοντας τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να διδαχθούμε ο ένας από την εμπειρία του άλλου. Είναι σημαντική φυσικά η παρακολούθηση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και να γίνεται μια διεθνή συνεργασία, γιατί το θέμα της ασφάλειας δεν είναι θέμα ενός κράτους μέλους μόνο. Βελτιώνοντας ε, και την ετοιμότητά μας, θα έχουμε την καλύτερη αντίδραση σε περίπτωση κατεπίγουσας κατάστασης. Επίσης, θα πρέπει να διδαχθούμε από τις εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει οι διάφορες χώρες με την μετάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Θα μπορούσαμε να συστήσουμε μια ομάδα με εμπειρογνώμονες και την 27 χωρών μελών προκειμένου να βοηθούμε σε αυτή τη διαδικασία και να καταρτήσουμε ίσως και μια βάση δεδομένων. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση για κάθε περίπτωση. Και στα μέτρα που θα προτείνουμε για την ασφάλεια, θα πρέπει να έχουμε υπόψη την ανάγκη αποτελεσματικότητας, αλλά και τις ορθολογικές δαπάνες. Ο Επίτροπος Έντιμπεργκ είχε επαφή με τις ε, πετρελαϊκές επιχειρήσεις για να ληφθούν κάποιες αποφάσεις ε, και να αποφύγουμε στη Βόρεια Θάλασσα παρόμοια φαινόμενα με αυτά που είχαμε με πετρελαιοκυλίδες. Θα πρέπει να ενεργήσουμε σε προκαταρκτική φάση, σε επίπεδο πρόληψης και, και όχι καταστολής, γιατί έτσι θα προστατεύσουμε καλύτερα τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φράνκο για το εξαιρετικό του έργο και συμφωνώ με όσα μόλις είπε ο συνάδελφος Ρούμπιχ. Πιστεύω ότι σωστά εμπνευστήκαμε από τις γνώσεις, τη σοφία, τη σύνεση που αξιοποιούμε πάντοτε στο έργο μας. Δηλαδή, ε, κοιτάζουμε τις καλές πρακτικές που ήδη υπάρχουν στις διάφορες χώρες, στα κυριότερα σημεία, κοιτάζουμε τι ισχύει στην πρακτική, στην πράξη μάλλον στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό προσυπογράφω και στο έργο του κυρίου Ρούμπιχ για τις διαβουλεύσεις με τους ε, πυρογνώμονες και τους ειδικού των ε, κρατών μελών. Πρέπει να δούμε πώς είναι διοργανωμένοι, πώς επιτελούν το έργο τους, τι απαντήσεις έχουν δώσει σε δύσκολες καταστάσεις όπου ενδεχομένω έχουν περιέλθει. Θα είχα να προσθέσω στα ζητήματα που εξετάσαμε μία και μόνη παρατήρηση. Θεωρώ ιδιαίτερα ευαίσθητο το θέμα και το γνωρίζω πλήρως ότι είναι πολύ ευαίσθητο, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να συζητηθεί και δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να καταφέρουμε να κάνουμε τροπολογίες, να υποβάλουμε τροπολογίες σχετικά. Θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντικό τον εξαιρετικό ρόλο που παίζει εδώ η ενημέρωση και από την αρνητική και από τη θετική της πλευρά. Ως προς τη θετική πλευρά σίγουρα είναι θεμελιώδου σημασία για όλο το έργο της πρόληψης, της γνώσης, για να ενημερώνεται διαρκώς ο πολίτης για τους κινδύνους που μπορεί να διατρέχει και για το ποια είναι τα μέσα που διαθέτει για να τους αντιμετωπίσει και ενδεχομένως να απειλήσει προβλήματα. Από την άλλη, και αυτό προκύπτει και από ένα επιχείρημα που ήδη αναφέρθηκε, την εμπειρία είχαμε με την επιδημία της γρήπης τον τελευταίο χειμώνα. Από την άλλη λοιπόν θεωρώ ότι η υπερβολική, υπέρμετρη ενημέρωση μπορεί στις επιμέρους χώρες, εδώ έχω απόψη τη δική μου χώρα αλλά φαντάζομαι συνέβη και σε άλλες χώρες, μπορεί λοιπόν να οδηγήσει σε μια κατάσταση ιδιαίτερης ανησυχίας μεταξύ των πολιτών. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να προκαλέσει και την απόφαση σε κρατικό επίπεδο να εξοπλιστούν με μια σειρά αποκρίσεων με ενδεχόμενες λύσεις που ήταν τελικά δυσανάλογες σε σχέση με, την... με τον μέγεθος του ίδιου του προβλήματος. Το καταλαβαίνω βέβαια και ακόμα και τώρα που το λέω γνωρίζω πως ευαίσθητο είναι το θέμα της ενημέρωσης, όμως πιθανώς θα ήταν καλό να συμπεριλάβουμε το στοιχείο αυτό μεταξύ των όσων θα συζητήσουμε μεταξύ μας στο διάλογό μας. Θα έπρεπε λοιπόν να βρούμε κάτι να πούμε και για αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις παρατηρήσεις και του Συγητού και του σκιώδου Συγητού, αλλά και των μελών της Επιτροπής σας. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκριθεί και υποβληθεί πριν από ένα χρόνο και στο μεταξύ υπήρξαν εξέλιξει. Το Συμβούλιο συμφώνησε για το σχέδιο δράση στα τέλη του προηγούμενου έτου. Πάντω, η συμβουλευτική ομάδα για το CBRN ήδη συγκροτήθηκε και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για μια ομάδα που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονε των κρατών μελών που επικουρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμβουλευτική ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Αλλά έχουμε κάποιες υποομάδες που εγκύπτουν σε συγκεκριμένες πτυχές του σχεδίου δράσης, πάλι με την βοήθεια των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών. Επίσης έχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες που μας επισήμαναν οι εμπειρογνώμονες. Και όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού φορέων. Αυτά λάβαμε υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που μας βρίσκουν σύμφωνος. Αυτά προς το παρόν, δεν έχω τίποτα άλλο. Καλώς σας ευχαριστούμε. Οπότε ολοκληρώσαμε το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Θα ψηφίσουμε, το... θα επανέλθουμε τον Ιούλιο στο θέμα αυτό. Οπότε, αφού ολοκληρώσουμε το σημείο 4, μπορούμε να επανέλθουμε στο σημείο 3 στο μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης και να δώσω το λόγο στον κύριο Κόφερ που θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις μια και αύριο θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Το σημείο αυτό που δεν φαίνονταν ιδιαίτερα ελκυστικό εξ αρχής, αρχίζει και γίνεται της μόδας πια. Σήμερα το πρωί είχαμε και μια δημόσια ακρόαση με θέμα το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική με εκπροσώπους ε, των διαφόρων φορέων του κλάδου, συμμετοχή της Επιτροπής ΙΜΚΟ και αναφέρθηκα με πάρα πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Είχα και πολλές συνομιλίες με συναδέλφους για το θέμα αυτό και η εντύπωση που αποκόμισα και τα συμπερέλαβα και στο κείμενο ε, Προφανώς όλα αυτά έτυχαν χάνει ενδιαφέροντος και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου ζητάτε ότι οι αρχές της, του ΠΟΕ πρέπει να τηρηθούν, δηλαδή ιδίω το θέμα της διαφάνειας. Αναφέρθηκε πλειστάκης πόσο σημαντικό είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να παίξουν τον σωστό και αρμόζοντα ρόλο. για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα προβλήματα είναι σε τρεις τομείς. Το κόστος, το περίπλοκο των προτύπων και το θέμα της συμμετοχής. Όσον αφορά το κόστος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν και συνενωμένα πρότυπα για, με μείωση των ε, τελών και επίσης να μπορεί κανένας να συμμετέχει online ε, σε μια συζήτηση να μην χρειάζεται δηλαδή, να πληρώνει για να μεταβαίνει κάπου για το ταξίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να προσθεθούν τα πρότυπα, ο αριθμός των ε, ε πιστοποιητικών παραδείγματος χάρη που απαιτείται να ε, μειωθεί. Τρίτον, θα ήθελα να αναφέρω ότι και στην ε, ακρόαση σήμερα το πρωί στην Επιτροπή ΙΜΚΟ δικαίως αναφέρθηκε ότι για τα πρότυπα η συνεργασία ε, με την έρευνα και ανάπτυξη ε, του ακαδημικού τομέα και του σχολικού τομέα είναι πάρα πολύ σημαντική. Η άλλη μου παρατήρηση είναι τεχνικής μορφής, πρόεδρος. Στο σημείο 10 τονίζω ότι θα ήταν καλό η Κομισιόν να προσπαθήσει να συντονίσει τις δραστηριότητες ε, τυποποίησης με τους ε, διεθνείς μας εταίρους. Ε, στο γερμανικό κείμενο αυτό το coordinate, το συντονίσω, δεν είναι νομίζω επαρκώς μεταφρασμένο. Ο όρος που χρησιμοποιείται στο γερμανικό κείμενο δεν είναι σωστό. Πρόεδρος, από ό,τι μου λένε διορθώθηκε ήδη το θέμα. Ο κ. Πανεγιάντοφ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπουτικόφερ, συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το προηγούμενο έργο του κυρίου Μπουτικόφερ. Οι προτάσει του θα βελτιώσουν τον τρόπο που η ευρωπαϊκή τυποποίηση λειτουργεί και έτσι καλωσορίζουμε τι προσπάθειέ του να γίνει αυτή η διαδικασία διαφανέστερη και πιο ανοιχτή η συμπερίληψη όλων των ενδιαφερομένων στη δικασία αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου μας. Για να διασφαλίσουμε κιόλα ότι και οι οργανώσεις των καταναλωτών θα μπορέσουν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί όταν, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των προτύπων. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή υλοποίηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προτύπων. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και κριτήρια επιλεξιμότητας για τους διάφορους φορείς. Και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ορθή ενημέρωση σε σχέση με τα πρότυπα και θα πρέπει να, να δούμε και τις δυνατότητες οργάνωσης ε, ενημερωτικών εξατιών. Η κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον ε, κύριο Μπουτικόφερ για την εξαιρετική του γνωμοδότηση και κυρίως και για την ακρόαση που διοργανώθηκε το πρωί στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Τέτοιου είδου εκδηλώσεις έπρεπε να οργανώνονται πολύ συχνότερα. Διότι δυστυχώς ε, οι δραστηριότητες τυποποίησης στην Ευρώπη δεν είναι αρκετά προβεβλημένες και γνωστές, ακόμη και αν πρόκειται για ένα στοιχείο θεμελιώδου σημασία και για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και για την εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι με την γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να βρούμε την ευκαιρία να, ρωτήσουμε, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισης της ανακοίνωσης που μας έχει υποσχεθεί. Πρόκειται για μια ανακοίνωση που αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης. Ένα σύστημα περισσότερο ολοκληρωμένο. Ένα σύστημα που αφορά συνολικά το πακέτο των μέτρων τυποποίησης και εδώ θα είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Ελπίζουμε στην ανακοίνωση λοιπόν να προσαρτηθεί και ένα πρόγραμμα δράσης όπου να αναφέρονται τα μέτρα αυτά και μεταξύ άλλων να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα προτύπων ενιαίο, πιο αποτελεσματικό, που να επιτρέπει πιο εύκολη πρόσβαση στα πρότυπα, ιδίως για τις κοινοτόμες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερα δυναμική δράση και έτσι να ενισχυθεί περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ρόλο της, στο σχεδιασμό προτύπων και στο διεθνές προσκήνιο. Και επίσης θέλουμε να υπάρχει και πιο βιώσιμη χρηματοδότηση στις δραστηριότητες τυποποίησης. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με τον κύριο Μπουτικόφερ όταν λέει ότι δυστυχώς το κόστος των προτύπων κάποιες φορές είναι ιδιαίτερα υψηλό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που όμως έχουν καινοτόμο δράση, πολύ καλές ιδέες, αλλά δεν έχουν τους πόρους, δεν έχουν έτσι πρόσβαση στα, πρότυπα. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι καθοριστική σημασία προφανώ και για το βιομηχανικό κλάδο, διότι ε, ενθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα και βοηθούν στην άρση των φραγμών στην αγορά. Έτσι όλοι γνωρίζουν και σέβονται τα πρότυπα που θεσπίζονται. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι είναι ζωτική σημασία να εξετάσουμε την ανακοίνωση Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της πρωινής ακρόασης, είδαμε ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, συνεργασία μεταξύ από τη μια των πανεπιστημιακών, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των ε, φορέων τυποποίησης της Ευρώπης. Θα έπρεπε και οι ακαδημαϊκοί να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία στις πρώτες φάσεις της για το σχεδιασμό των προτύπων. Θεωρώ λοιπόν ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να ενημερώνεται συστηματικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εντολή που ανατίθεται από καιρού καιρών για την διαδικασία τυποποίηση, είτε είναι ετήσια είτε διετή. Την εντολή αυτή την εκχωρεί η Επιτροπή και αφορά τι δραστηριότητε τυποποίηση και τη χρηματοδότησή του. Για άλλη μια φορά λοιπόν, συγχαρητήρια στον κύριο Μπουτικόφερ θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες, όμως οι τροπολογίες αυτές στόχο θα έχουν απλώς να, εμπλωτί, να εμπλουτίσουν το κείμενο και να εδρεώσουν τον χαρακτήρα της τυποποίησης, όπως ήδη περιγράφεται. Ε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ χαίρομαι που η συζήτηση έχει ξεκινήσει τώρα. Γιατί η τυποποίηση όπως και το θέμα των ε, ε, <clears throat> ευρυστεχνιών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδίως γιατί έτσι εκμεταλλεύονται τις ε, τεχνολογικές γνώσεις που βασίζονται στην τυποποίηση και που καλύπτονται και από πολλές καινοτομίες. Αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα είναι το κύριο πρόβλημα του να εξεύρουμε δηλαδή τα σωστά πρότυπα. Θα πρέπει από πλευράς Κομισιόν να σκεφτούμε πως στο μέλλον θα καθορίσουμε τα πρότυπα με τέτοιο τρόπο τους ώστε να είναι εύκολη η αναζήτησή τους ε, στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες περιλήψεις abstracts που θα πρέπει να είναι κατά δυνατόν πολύγλωσσες, ε, ούτως ώστε σε όλη την Ευρώπη να μπορεί κανένας να διαβάσει αυτά τα κείμενα. Η δεύτερη μου παρατηρήση αφορά την ε, δομή της οργάνωσης αυτής ε, ε, τυποποίησης. Ίσως θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο πρότυπο ή ένα νομικό πλαίσιο της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου Βέβαια και των Ορμοδίων Υπουργών μετά από την ε, ανακοίνωση αυτή θα είναι θέμα σημαντικό η πιστοποίηση αυτών των ε, Ινστιτούτων ε, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα. εάν ε, κάτι αναγνωρίζεται παραδείγματος χάρη ένα κράτος μέλος, αναρωτηθεί και στο άλλο. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η αμοιβαία αναγνώριση. Αυτό θα ήταν μια ε, δυνατότητα. Απ' την άλλη μεριά, οι υπηρεσίε τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ασχολούνται με την εναρμόνιση, ούτως ώστε θα ήταν δυνατόν να υπάρχουν και ανταγωνιστικά συστήματα. Όταν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούν να ενσωματωθούν στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο συνάδελφος Λάνε. Äh, Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό που είπε η συνάδελφος Τίκαου. Κύριε Μπιουτικόφερ, ίσως θα έπρεπε να ε, πούμε στην Κομισιόν το θέμα του ότι θα πρέπει γλίγορα να υποβάλει μια γενική μεταρρύθμιση του συστήματος τυποποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα τα οποία και εσείς θίξατε, που απαιτούν γενικής ε, μεταρρύθμισης και εκεί θα πρέπει να ασκήσουμε νομισοποίηση για να μπορέσει η Κομισιόν να ξεκινήσει και να προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Αφενός το θέμα είναι πώς μπορούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα να το τοποθετήσουμε στο παγκοσμιοποιημένο πεδίο τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και τη βιομηχανία μας, θα πρέπει να επιταχύνουμε επίσης τη διαδικασία τυποποίησης και όσον αφορά την χορήγηση της εντολής θα πρέπει να το σκεφτούμε επίσης, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε τεχνολογικές ε, καινοτομίες που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πρότυπα. Παραδείγματος χάρη συζητάμε το θέμα της ε, ηλεκτρικής κινητικότητας και βλέπουμε πόσο πόσο καθυστερούμε εδώ από το θέμα της πρίζας που χρησιμοποιείται και πέρα. Λοιπόν, εδώ πάλι είναι το θέμα της ε, χορήγησης της εντολής, ούτως ώστε τα πρότυπα αυτά να εφαρμόζονται γρήγορα. Θα πρέπει και αυτό να το σε αυτή τη δέσμη. Και έχω και μια ξεκάθαρη ερώτηση για το κόστος. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το σύστημα είναι πολύπλοκο βέβαια. Αλλά δεν ξέρω για το κόστος κατά πόσο είναι τόσο μεγάλο το εμπόδιο. Εάν έχω ενημερωθεί σωστά, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, θα πρέπει να ορίζονται κατά κάποιο τρόπο πρότυπα με κάποια χίλια, χίλια ευρώ. Όταν κανένας όμως είναι ο πρόσωπος που υποβάλλει ένα πρότυπο έχει και ένα οικονομικό όφελος. Είναι λοιπόν πραγματικά τόσο μεγάλο το, το πρόβλημα το κόστος. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Καλή ερώτηση. κυρία Σαρτόρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμμεριστώ το μεγαλύτερο μέρος του στι παρεμβάσει των συναδέλφων. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή τη αρχική φάση των διαβουλεύσεων και συζητήσεων, διότι το φθινόπωρο προβλέπεται μάλλον μια σειρά από εκθέσει και εισηγήσει που αφορούν ακριβώ αυτό το θέμα και στην ε, δική μας την Επιτροπή και στην Επιτροπή της Ιστορικής Αγοράς. Νομίζω ότι η βασική μέρημνα που θέλουμε να καλύψουμε, μέρημνα που αντικατοπτρίζονται στις προτάσεις του συναδέλφου, είναι το κόστος, όπως ανέφερε και ο τελευταίος συνάδελφος, αλλά ακόμη όταν ιδίω μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η δυσκολία που έχουν οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν πρόσβαση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επειδή εκεί συνεχώς νέα βάρη που και νέες υποχρεώσεις πρέπει να σεβαστούν, νέο κόστος λοιπόν. Ένα, μια λύση λοιπόν που θα υποχρέωνε με τρόπο σαφή να απλουστευθούν τα πρότυπα είναι ένας στόχος ακριβώς που θα πρέπει να επιδιώξουμε. Οι προτάσεις λοιπόν αυτές θα πρέπει να μας οδηγήσουν και στο εξής συμπέρασμα. Προφανώς ε, η πρόσκληση της Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτη να συντονίσουμε τις δραστηριότητες τυποποίησης με τους ε, συνομιλητές και τους φορείς τους διεθνείς, ιδιαίτερα με τις Ηνωμένε Πολιτείες, διότι αυτό θα πρέπει να γίνει κανόνας πρότυπο, λέει η για όσα θα γίνουν από σήμερα και στο μέλλον. Η Ευρώπη θα πρέπει συνεχώς να εξετάζει τους νέους κανόνες, τις νέες, τα νέα πρότυπα που βλέπονται και στις άλλες χώρες. Διότι ανάλογα με το τι γίνεται στις άλλες χώρες, τότε και οι δικοί μας συνομιλητές με τους συνομιλητές μας μάλλον, θα καταλαβαίνουμε κατά πόσον θα αφορούν τα δικά τους τα μέτρα τις δικές μας τις ε, βιομηχανίες, το μηχανικό κλάδο. Θα πρέπει λοιπόν κάθε φορά να διαλέγουμε μεταξύ των στοιχείων που θα καθιστούν σκόπιμη ή όχι τη μια ή την άλλη επιλογή. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα τον συνάδελφο και ελπίζω να ακολουθούμε στο μέλλον διαρκώς τον κανόνα αυτό, που κάποτε παλιότερα τον ακολουθούσαμε και κάποτε όχι. Euh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Μπιουτικόφερ. Euh- Γιατί ήταν ε, πολύ σωστή διαδικασία που εφάρμοσε και που κατέληξε στην έκθεση αυτή. Οι κανόνες αυτοί και τα πρότυπα αυτά ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προέρχονται από τρίτη χώρες. Πρόκειται για προϊόντα και υπηρεσίες εισαγωγή Και από αυτή την άποψη τα πρότυπα αυτά συνιστούν ένα είδο προστασίας για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Αυτό που θα ήθελα να πω, πέραν αυτών που ανέφεραν οι προλαλήσαντες, ίσως δεν έχει άμεση σχέση με την έκθεση του κ. Μπουτικόφερ, που επικεντρώνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ αφορά τους ελέγχους τα σώματα ελέγχου και τις ε, ελεγκτικές διαδικασίες, γιατί μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε τους κανονισμούς, τις ρυθμίσεις και τους κανόνες, αλλά τα σώματα των ελεγκτικών διαδικασίες ελέγχου αυτή τη στιγμή είναι ανεπαρκή στην Ευρώπη. Και αυτό φαίνεται όταν το συγκρίνουμε με τους ομολόγους μας είτε των Ηνωμένων Πολιτειών είτε των αναδειωμένων οικονομιών. Γιατί έχουμε εμεί κάποιου κανόνε και πρότυπα, αλλά δεν ξέρουμε αν γίνονται σεβαστά. Γιατί δεν υπάρχουν αρκετέ ελεκτικέ διαδικασίε ή αρκετοί ελεκτέ για να εξακριβώσουν την εφαρμογή του. Πέραν τη κανονιστική και ρυθμιστική δραστηριότητα που είναι πλούσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό θα ήταν να εγγύψουμε και στο θέμα των ελέγχων. Ποιε είναι οι ελεκτικέ διαδικασίε και ποια είναι τα σώματα ελεκτών για ελέγχου που υπάρχουν στην Ευρώπη που εξασφαλίζουν την ε, σωστή εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται στην Ευρώπη, αλλά και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εισάγουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ στον Φωσπιτικόφερ πάλι και μετά η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συμβολή τους. Θα ήθελα να αναφερθώ σε λίγα από τα ερωτήματα που υποβληθούν. Η κυρία Βάσενχομ, η αρμόδια αντιμετάρχη στην Κομισιόν, στη Γενική Διεύθυνση Enterprise επιχειρήσεων, τόνισε σήμερα το πρωί ότι η Κομισιόν προτείνεται το φθινόπωρο ή αρχές του έτους, ο κύριος ε, Ταγιάννη είπε στα τέλη του έτους, να υποβάλει μία δέσμη μέτρων για την τυποποίηση θα ξεπερνάει οπωσδήποτε αυτά που υπάρχουν εδώ στην γνωμοδότηση. Είναι πολύ πιο ευρύ. Και όταν έχουμε αυτή τη δέσμη, κυρία Λάγκε, θα μπορέσουμε να σκεφτούμε κατά πόσον είναι επαρκές ή όχι. Ε, θα υπάρχει βέβαια και η πρωτοβουλία του συνάδελφου Ζούστρικ από τη Τσεχία που έχει σαν στόχο να δώσει κάποιες συμβολές ε, Τώρα το κόστος, κατά πόσο αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα, δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Αλλά παραδείγματο χάρη έχοντα ακούσει αυτό που είπε ο Κουτσογιάννη, είναι ένα από τα πολλά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι το θέμα τη συμμετοχή. Σε ορισμένα κράτη-μέλη οι ΜΜΕ συμμετέχουν πολύ καλά, σε άλλε λιγότερο. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της πρόσβασης στα πρότυπα. Ε, να μπορούμε να κατανοηθούν τα πρότυπα αυτά. Είπε κάποια σχετικά πράγματα εδώ ο κύριος Ρούμπικ. Και μετά είναι το πρόβλημα του κόστους. Και το θέμα δεν είναι ότι όλα τα πρότυπα θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν. Αυτό θα κατέστρεφε και κάποια επιχειρησιακά πρότυπα που είναι λογικά. Αλλά παραδείγματο χάνει στην οργάνωση DIN υπάρχουν κάποιες προσφορές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια δέσμη δηλαδή προτύπων με χαμηλό τέλος και αυτό είναι πολύ ευνοϊκό. Και μετά και μια απλούστευση της διαδικασίας. Αυτό είναι αυτό που είναι δυνατόν να γίνει για τις ΜΜΕ. Το κόστος δηλαδή παίζει κάποιο ρόλο, χωρίς να είναι καθοριστικό. Η κυρία είναι από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Μπιουτικόφερ ότι οι δέσμοι τυποποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι έτοιμοι από στιγμή σε στιγμή και στην ανακοίνωση θα προβλέψουμε ε, κάποιες δράσεις και ένα νομοθετικό πλαίσιο για το τέλη του έτους. Από ό,τι κατάλαβα, εσείς παροτρύνετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει άμεση δράση, αλλά είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία γιατί ζητάμε κάτι καινούριο από την τυποποίηση. Ζητούμε τυποποίηση, αλλά σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και υπάρχει ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο. Και έχουμε μεν εναρμονισμένα πρότυπα, αλλά έχουμε και μια νέα προσέγγιση. Και ξαφνικά λέμε ότι θέλουμε συνεργασία με, την, με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Τυποποίησης για να ληφθεί υπόψη και η καινοτομία. Και αυτό είναι μια νέα προσέγγιση, οπότε θα πρέπει να αλλάξουν πολλές διαδικασίες. Θα το σκεφτούμε λοιπόν και αυτό και φυσικά θα πρέπει η νέα προσέγγιση ε, να γίνει κατανοητή, να τύχει συμφωνίας και να δούμε και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούμε και να τους δοκιμάσουμε πριν γίνουν ρηξικέλευτες αναθεωρίες γιατί αυτή τη στιγμή η διαδικασία τυποποίησης λειτουργεί σωστά. Ας είμαστε προσεκτικοί λοιπόν να μην καταστρέψουμε τα θετικά στοιχεία της. Επίσης ζητούμε κάτι καινούριο παραλαμβάνω. Ζητούμε από τις αρμόδιες για την τυποποίηση αρχές να κάνουν κάτι σε συνεργασία με την κοινοτική νομοθεσία, το κοινοτικό δίκαιο και από εκεί θα προκύψουν νέες προκλήσεις. Και θα αρχίσουν όλες αυτές τις συζητήσεις τώρα, αλλά είναι μια διαδικασία που θα γίνει από τη βάση προς τα πάνω, σε συνεργασία με τις αρχές τυποποίησης και σε συνεργασία με τις επιχειρίες. Γιατί δεν είναι μία διαδικασία που ενορχιστρώνει και εκτελεί μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά γίνεται σε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τις αρχές τυποποίησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι αύριο πέντε απόγευμα είναι η λήξη της προθεσμίας για τις τροπολογίες. Ασυνήθιστο, αλλά έχει συμφωνηθεί. Και σας παρακαλώ να τηρήσετε αυτή την προθεσμία για να μπορέσουμε να ε, προφτάσουμε να ετοιμάσουμε τις μεταφράσεις του κειμένου κλπ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν εδώ την εξάρτηση αυτού του σημείου της διάταξης και ολοκληρώνουμε και τη συνεδρίαση και μπορείτε να πάτε σε άλλες συνεδριάσεις τώρα. Μόνο οι συνάδελφοι συντονιστές θα παραμείνουμε εδώ γιατί θα αρχίσουμε αμέσως με τις συνεδριάσεις των συντονιστών.